Very good. Uh, Καλό απόγευμα και πάλι. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίασή μα μετά από αυτή τη μικρή διακοπή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να χαιρετήσω για τελευταία φορά σε αυτή τη θητεία το Μισελ Μπαρνιά στην Επιτροπή Εσωτερική Αγορά. Είναι ο Επίτροπο, ο οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα εσωτερική αγορά και τι υπηρεσίε τη εσωτερική αγορά. Είναι πραγματικά ήταν τιμή και προνόμιο για μας να τον υποδεχτούμε πολλές φορές στην Επιτροπή μας μετά από την ανάληψη καθηκόντων τους. Αλλά θυμάμαι ότι ήσασταν και μέλος της Επιτροπής μας και ενεργός βουλευτής, έστω για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και ποιος ξέρει μπορεί να θέλετε να επανέλθετε στην Επιτροπή αυτή στο μέλλον. Είναι πολύ χρήσιμο πάντως που είναι τόσο πολλοί βουλευτές εδώ παρόντες. Θα δώσω το λόγο σε λίγο στον Μισελ Μπαρνιέ για να μας μιλήσει για τις σκέψεις του σε σχέση με τη συνεργασία μας και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Έχουμε όμως μερικά σημαντικά επιτεύγματα τα οποία μπορούμε να εξάρουμε, ιδιαίτερα του, την νομοθεσία για την ενία αγορά. Φυσικά παραμένουν και πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο μέλλον και σίγουρα ο Μισελ Μπαρνιέ θα αναφερθεί στο ρόλο μας και θα αναφερθεί και στα θέματα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς και τα άλλα σημαντικά ζητήματα ενώπιών μας για το μέλλον. Ε, κανονικά προβλεπόταν να τελειώσουμε στις 6 και 10. Βλέπω κάτι μπουκάλια και κάτι ποτήρια να ετοιμάζονται έξω από την αίθουσα. Ίσως αυτό σας παροτρύνει να είσαστε σε πιο σύντομη ερωτήσει, σα, γιατί αλλιώς θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο στο κοκτέιλ. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω διατυπώσει, θα ήθελα να δώσω αμέσω το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ, τον Μισελ, να λάβει το λόγο και μετά όποιο θέλει μπορεί να ζητήσει να εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών. Ο πάνω θα καταγράφει του ε, ομιλητέ. και με μεγάλη χαρά λοιπόν έδωσε στον Μισελ Μπαρνιέ το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνάντηση που κάνουμε σήμερα γύρω από αυτή τη στρογγυλή τράπεζα εξάλλου. Δεν είναι καθημερινό αυτό, αλλά και αυτό είναι πολύ θετικό σε σχέση με το πνεύμα το οποίο πάντα ε, διέπνε τις συναντήσεις μας τα τελευταία χρόνια. Μια στρογγυλή τράπεζα όπου ο καθένας βρίσκει τη θέση του, όπου υπάρχει εγκαρδιότητα, υπάρχει συμβολισμός λοιπόν το ότι όλοι είμαστε γύρω από ένα κοινό στρογγυλό τραπέζι και αυτό αντανακλά και το ε, επικοδομητικό και φιλικό πνεύμα το οποίο επικράτησε στις ε, συναντήσεις μας και στην εργασία μας. Η εργασία μας δεν ήταν πάντα καθαρά θεσμικού χαρακτήρα, δεν ήταν κλασικά θεσμική και μόνο, αλλά υπήρξε ένα κοινό πνεύμα που μας ένωνε όλους μας και εφόσον είναι και η τελευταία φορά που γίνεται αυτή η συνάντηση, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το πνεύμα, ο καθένας από εσά, αλλά και οι συνεργάτες σας, οι οποίοι και αυτοί έχουν συνεργαστεί μαζί σας σε τόσες εκθέσεις, όλη η γραμματεία της Επιτροπής που υποστήριξε τον Μάλκον, και εγώ γνώρισα αυτή την Επιτροπή ως ένας από εσά, ως μέλος της Επιτροπής για κάποιους μήνες, πάντα ένιωθα μεγάλη ε, έκπληξη, αν θέλετε, εντυπωσιαζόμουν από τον τεράστιο αριθμό των θεμάτων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και όταν ανέλαβα το έργο του Επιτρόπου, σίγουρα είχα πάντα την υποστήριξη και τη βοήθεια της Επιτροπής σας και της Γραμματείας της Επιτροπής σας για την πολύ καλή συνεργασία και το πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας. Δεν ξέρω λοιπόν πώς να το πω αυτό, πόσο μέτρησε αυτό το επικοδομητικό πνεύμα για να μπορέσω να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις που όπως θυμόσαστε είχα αναλάβει στην ε, ακρόασή μου πριν από την αναλέψη καθηκόντων ενώπιον της κοινή συνεδρίασης των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΙΜΚΟ. Μέσα στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν αυτή την ακρόαση προσπάθησα να εξασφαλίσω την συμφιλίωση κατά κάποιο τρόπο των πολιτών και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την ενιαία αγορά. Γιατί όλοι αυτοί είχαν την εντύπωση ότι η ενιαία αγορά ήταν ένα εγχείρημα προς όφελος των μεγάλων εταιριών και δεν τους αφορούσε. Ενώ με την ενιαία αγορά μπορέσαμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων υπήρχε μια δυσπιστία και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο και του ευρωσκεπτικισμού πολλές φορές. Γι' αυτό θα ήθελα με κάποιο προδραστικό τρόπο να κάνω ένα απολογισμό του τι έχουμε κάνει, αλλά θέλω να τονίσω ότι η προσήλωσή μας στην προσπάθεια συμφιλίωση των πολιτών με την εσωτερική αγορά ήταν κάτι το οποίο προχώρησε και εξάλλου χάρη στο γεγονό και ότι η Επιτροπή σας Μάλκον δεν περίμενε τι προτάσει τη Κομισιόν, Πολλέ φορέ με εκθέσει πρωτοβουλία ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, εκθέσει πρωτοβουλία που ήταν πάρα πολύ χρήσιμε και οι οποίε επέτρεψαν να γίνει σαφής η θέση και οι αιτήσει των ε, επαγγελματιών, των πολιτών, των τοπικών εκλεγμένων κτλ. Είναι πάρα πολλέ λοιπόν οι πρωτοβουλίε που αναλάβαμε μαζί για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίω το πρώτο φόρουμ τη ενιαία αγορά το οποίο έλαβε χώρα στην Κρακοβία, μετά η εβδομάδα τη ενιαία αγορά, ο μήνα τη ενιαία αγορά. Και με τον τρόπο αυτό ανοίξαμε διάπλατα πόρτες και παράθυρα στην ενιαία αγορά, ώστε να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να το κατανοήσουν και η Επιτροπή σας ήταν πάντα ένας εταίρος για μένα και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την βοήθειά σας, όπως ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και τον Μάλκον Χάρμπορ, γιατί είχα την ευκαιρία να εργαστώ υπό την ηγεσία του, που ήταν μια ηγεσία εξαιρετικά ικανή, επακριβής, ποτέ χαλαρή, πάντα επικοδομητική. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Τι θέλουμε να κάνουμε μαζί. για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά την εσωτερική, την ενιαία αγορά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να εξηγήσουμε ότι είναι πράγματι ένα ατού, ένας μοχλός εξόδου από την κρίση. Ένας μοχλός ανάπτυξης, αλλά και ένας χώρος όπου μπορεί να υπάρχει και να πάλεται μια κοινή οικονομική ζωή. Και υπενθυμίζω ότι πριν από πέντε χρόνια είχε παρουσιάσει ο Μάριο Μόντι την λεγόμενη διάγνωση για την κόπωση της εσωτερικής αγοράς, μια πολύ σημαντική έκθεση επίσης του συναδέλφου σας του Λουί είχε εκφράσει ακριβώς την απόσταση που χωρίζει την εσωτερική αγορά από τους πολίτες, την κόπωση αυτή και φυσικά ο κίνδυνος κρίσης από την οποία δεν έχουμε εξέλθει πλήρως μπορεί να οδηγήσει και πάλι σε εθνικές αναδιπλώσεις, ακόμα και εθνικιστικές μορφές ε, αναδίπλωσης που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο οικονομικό προστατευτισμό. Ο καθένα για τον εαυτό του, ο καθένα στο δικό του παχνί. Γι' αυτό εγώ ενθαρρύνθηκα ιδιαίτερα από την προσπάθεια της δικής σας Επιτροπής να δημιουργήσουμε, να προετοιμάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο σε εσά που το βαφτίσατε, ονομάσαμε πράξη, πράξεις για την ενιαία αγορά, μία σειρά από πρωτοβουλίε, υπήρξε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά τέτοιων πρωτοβουλειών, ελπίζουμε θα υπάρξει και τρίτη, Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν κυρίως τέσσερα θέματα τα οποία μπορέσαμε να προχωρήσουμε χάρη σε εσά και με εσά. Η μεταρρύθμιση των δημοσίων προμηθειών πρώτα, για να μπορεί να απλοποιηθεί και να γίνει με πιο στοχευμένο τρόπο, γιατί είναι το 18% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για ως μοχλός ανάπτυξης το σύνολο των δημοσίων προμηθειών να έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και το πιο ισοδίκαιο χαρακτήρα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάρκ Ταραμπέλα και τον Φιλίπ Ζουβάν, αλλά και τον πρόεδρο Χάρμπο και όλου από εσά οι οποίοι συνέβαλαν και είναι πολλοί από εσά μέσα σε αυτή την αίθουσα που υπήρξαν σκιώδει συζητητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων που όλα αυτά μα επέτρεψαν να δημιουργήσουμε ένα νέο κόρπου κανόνων πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο απλοποιημένο και πιο ασφαλές και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας επιλογής για τα κράτη και τις τοπικές αρχές και τους κοινού ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε πρόκειται για δημόσιες ε, προμήθειες αγαθών, είτε για παραχωρήσεις, συμβάσεις παραχωρήσεων. Επίσης το θέμα της αϊλοποίησης των τιμολογίων στο δημόσιο τομέα ήταν η έκθεση Λάγκεν και άλλων που ουσιαστικά υλοποιήθηκε σε ένα χρόνο ρεκόρ και οδήγησε στην αϊλοποίηση των διαδικασιών όπως προβλέπεται από την αρμόδια οδηγία. Και σας υπενθυμίζω ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το e-invoicing, θα επιτρέψει εξοικονομήσεις της τάξης των 2 δισεκατομμύριων ευρώ το χρόνο. Και ερχόμαστε εδώ στο θέμα της ψηφιοποίησης, της αποϊλοποίησης των δημοσίων λογαριασμών και θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν χρειαζόμαστε τόσο δημόσιο χρήμα και τόσο ιδιωτικό χρήμα για να επενδύσουμε στην καινοτομία, ότι αν πετύχουμε το στόχο αυτό να μην χρειάζεται πια υποστήριξη σε χαρτί όλων αυτών των λογαριασμών, θα εξοικονομήσουμε 80 δισεκατομμύρια το μήνα σε, ε, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους, ε, σε άλλους τομείς. και δεν αναφέρθηκα στο θεσμικό πλαίσιο πλήρως για τις δημόσιες ε, αγορές που θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί εκεί πέρα μια συμβαστική λύση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο θέμα. Ένα δεύτερο μεγάλο, ένας δεύτερος μεγάλος τομέας ήταν οι υπηρεσίες και γνωρίζετε πολύ καλά την ε, οδηγία για τις ε, υπηρεσίες που οδήγησε σε τόσες συζητήσεις και διαμάχες φυσικά τώρα έχουν ε, ηρεμήσει τα πράγματα αλλά δεν πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί ως μια επιταγή των Βρυξελών, κάτι το οποίο γίνεται εκ των άνω, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη. Να υπάρχουν και πρωτοβουλίες εκ των κάτω. Έχουμε πολλές εδώ πρωτοβουλίες, όπως ήταν η οδηγία για τις υπηρεσίες όπου έχουμε περάσει πολλούς κοπέλους και έχουμε περάσει πολλές δύσκολες καμπές ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια σημαντική πολιτική όθηση για αυτό το ε, κείμενο και εδώ πρέπει να τονίσω και τη σημασία του Ανδρέας Βάπ, της Μαρία Κοράτσαμπίλ και πολλών άλλων. Μπορέσαμε να δώσουμε λοιπόν μια νέα πολιτική όθηση στο κείμενο αυτό υπογραμμίζοντας τη σημασία του να υπάρξει μια οικονομία υπηρεσιών μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομική ζωή. Η μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την μη εφαρμογή και μεταγραφή των ε, οδηγιών. Εδώ δεν υπήρξε λοιπόν καμία παρέκκληση από την ε, Κομισιόν. Ήμασταν απόλυτα σαφείς για το θέμα αυτό και πολύ αυστηροί. Συμφωνήσαμε να μην αναθεωρήσουμε αυτό το κείμενο για τις ε, υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε για εφαρμόζοντας αυτό το, το κείμενο και όχι αλλάζοντας το όπως ζήτησαν ορισμένοι Βρετανοί συνάδελφοι που θεωρούσαν δεν προχωράει αρκετά και έτσι μπορέσαμε να βελτιώσουμε τους κανόνες της καθημερινής ζωής και να κάνουμε αυτή την οδηγία πιο φιλική προς το χρήστη με μεγαλύτερη ε, διευθύνση του ρόλου του τελικού καταναλωτή προς τον οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες και με πρακτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ασφάλισής τους που ήταν πολλές φορές πολύ αν, ανώμια στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο, πολλοί από εσά που ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά πρέπει να συνεχίσουν αυτό το εγχείρημα και να αποφύγουν ότι θα επανέλθει μια περίοδος κόπωση σε σχέση με αυτή την οδηγία. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω το έργο του Μπερνάντε Βερνιό και της ε, Κωνστάνς και άλλων, της Χάιντι Ρούλε, του Τόμας Χέντελ, για τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι ένα κείμενο που απευθύνεται στους πολίτες, πάρα πολύ συγκεκριμένο, που ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη και που πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και της κινητικότητας. Νομίζω ότι εργαστήκαμε πολύ καλά από κοινού για να υποστηρίξουμε τους ε, επαγγελματίες οι οποίοι πρέπει να μετακινούνται από μια χώρα στην άλλη διευκολύναμε τις διαδικασίες και επίσης χάρη στην ε, Ευρωπαϊκή Κάρτα και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες έχουμε επιταχύνει ιδιαίτερα την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι βρήκαμε μια σωστή ε, ισορροπία σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα προσόντα, την προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλες χώρες, την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Προσόντων και του Μηχανισμού Προειδοποίησης για τα θέματα ασφάλειας των ασθενών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος όλων αυτών των νέων ρυθμίσεων στην πράξη και να τις αξιολογήσουμε, να ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια και αμοιβαία αξιολόγηση, να δούμε καλύτερα τα επαγγέλματα τα οποία διέπονται από ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλέγμα και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα. Για τον τομέα των υπηρεσιών επίση θέλω να αναφερθώ για στι πρωτοβουλίε όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή σα και όπου η Επιτροπή σα έχει δώσει την άποψή τη, έχει πολλέ φορέ κρατήσει και μια κριτική στάση. Πρόκειται καταρχήν για τι πρακτικέ που έχουν να κάνουν τα στεγαστικά δάνεια με την συμβολή του Κουρτ Λέχνερ την πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό για όλου. κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλου. όπου που ο κύριος ε, Κλούτε ήταν εισηγητής σε μια άλλη επιτροπή ε, και η κυρία Λίνκεμπα και επίσης η κατάρτιση των ε, καταναλωτών σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα με τον κύριο Παντσέρη. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό συζήτησα τα θέματα φυσικά και με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν προκτελεί μόνο για τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, του φορεί πιστοληπτικής αξιολόγησης. Δεν είναι μόνο αυτά. Η οικονομία πρέπει και οι πολίτες να είναι καλύτερα ε, πληροφορημένοι. 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είχαν τύχει, είχαν προσκούσει σε άρνηση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού τα τελευταία χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό η ενιαία αγορά υπηρεσιών και η ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες. Ένας τρίτος σημαντικός χώρος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίω η υποστήριξη στις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό το έκανα με τη βοήθεια του συναδέλφου μου επιτρόπου του κυρίου Ταγιανή, μια νέα προσέγγιση για το κεφαλαίο για την πρόσβαση σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερη έμφαση που δώσαμε για το Ταμείο ε, Κεφαλογικών ε, Αποθεμάτων και Επαρχιών που είναι απαραίτητο για να μειώσουμε το βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δυνατότητες για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας χρηματοδότηση που θα το αντιμετωπίσουμε και στην επόμενη θητεία και επίσης να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα της ε, νέας οικονομίας όπως λέγεται το οποίο πρέπει να σας ενδιαφέρει, τους νέους τρόπους του λεγόμενου crowdfunding, της ε, μαζικής χρηματοδότησης από πολλούς μικρούς επενδυτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάστηκε στην, ε, ε, στην έκθεση που παρουσίασε, ο λεγόμενος πληθοπορισμός. Πολλές φορές έχετε λοιπόν καταστάσεις όπου υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτήν την μορφή μαζικής χρηματοδότησης πληθοπορισμού και αυτό σε τομείς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όπως είναι η γεωργία ή τα πολιτιστικά θέματα. Έχουμε ε, αντιμετωπίσει το θέμα του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας και εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα αγαπητοί κύριοι βουλευτές από την επιτυχία μια συνδιάσκεψη που οργάνωσα με τον κύριο Ταγιάννη μαζί και με παρουσία πολλών από εσά στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο. Ήταν 2.000 άτομα πολλές μέρες κιόλα, χωρίς να υπάρχουν απλώς μονόλογοι, ήταν σε πολλά εργαστήρια συμμετοχικού. Και πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία αλλάζουν σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει εμείς να είμαστε ιδιαίτερα ευήκοοι και να ενδιαφερόμαστε για αυτήν την ανάδυση νέων μορφών επιχειρήν και νέων επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων πολλές φορές. Αυτό ήταν και ο στόχος αυτού του, αυτής της συνδιάσκεψης για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική κ. Ταραμπέλα ήταν εδώ οι παρόν και πολλοί άλλοι, για να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα προβλήματα της κοινωνικής οικονομίας. Τέταρτος χώρος επίσης, η, προσ... η προσαρμογή της ενίας αγοράς για ε, ενώπιον των ψηφιακών προκλήσεων. Εκεί συνεργαστήκαμε και με την κυρία Κρούζ, ώστε η ενία αγορά να μπορέσει να είναι επίκαιρη να ζει στον 21ο αιώνα, που είναι ο αιώνα ο αιωνας ολη τη Ευρώπη, να μπορεί να λάβει υπόψη την παρουσία του διαδικτύου και τις, ε, να λάβει υπόψη τις αιτήσει των πολιτών και των καταναλωτών. Ο ρυθμός της ε, κοινοτομία είναι πολύ γρήγορο και είναι πιο γρήγορο από το ρυθμό τη νομοθεσία. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά χάρη στη δική σα υποστήριξη μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε ένα θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που έχει προοδευτικό χαρακτήρα μέχρι το 2015-2020. Συζητήσαμε με του εμπλεκομένου πριν από δύο χρόνια και είχα προτείνει ένα σχέδιο δράση για να μπορέσουμε να άρουμε τα εμπόδια για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιγραμμικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τι εργασίε οι οποίε έγιναν από τον Άριο Σεβαριά, τον κύριο Κατάινεν, τον κύριο Κουρέιντ Κάμψ και σε δύο από αυτέ τι συνεδριάσει που είχατε διοργανώσει είχα εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από την ικανότητά σας και το ενδιαφέρον σας για αυτές τις ενέργειες. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ε, επιγραμμικές υπηρεσίες ε, τα, πάνω από τα τρία τέταρτα της δουλειάς αυτής έχουν ήδη εφαρμοστεί για την προστασία των καταναλωτών, για την οδηγία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ε, για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, για τα sites συγκριτικής παρουσίασης τιμών και την προστασία των δεδομένων. Τρία ακόμη κείμενα θα ήθελα να σας παρουσιάσω που έχουν δρομολογηθεί για την εσωτερική αγορά, το θέμα του Αρίας για την παράδοση δεμάτων ε, ο κύριος Κρόιτσμαν, ε, η κυρία Ρούλε και πολλοί άλλοι, η κυρία Μπιέλαν ε, επίσης, εργάστηκαν επ' αυτού και είναι ένα πραγματικό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί μεταξύ κρατών μελών για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο σε σχέση πάντοτε με την προστασία των καταναλωτών. Όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, σαλιδεμόζε, Φόξ, Ρούλε, Ντε Ιούγκ, όλοι εργάστηκαν ε, για να ε, υπάρξουν μέτρα πλαισίωσης ε, των τυχερών παιχνιδιών χωρίς να εισαχθούν νέα μέσα ή νέα νομοθετικά κείμενα όσον αφορά το θέμα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ένα θέμα πολύ σημαντικό, ακόμη κι αν ε, επισήμως η δική σας Επιτροπή δεν πραγματεύεται το θέμα αυτό, το πακέτο των πληρωμών είναι ε, ε, τμήμα αναπόσπαστο της δουλειάς μας. Την Πέμπτη στην Ολομέλεια ε, ελήφθησαν αποφάσεις που θα συνοδεύσουν τη δουλειά μας στην επόμενη θητεία. Καταρχάς, ε, χάρηκα πάρα πολύ που ήταν επιτυχημένες ε, οι διασκέψεις ε, του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου για τα επαγγελματικά προσόντα, ε, γιατί μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, να δούμε πώς εφαρμόστηκαν στην πράξη αυτά τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στα κείμενά μας. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες να ε, ξαναρχίσει πάλι μια συζήτηση τη στιγμή της εφαρμογής των ε, ε, κειμένων αυτών. Ας μην υπερβάλλουμε όμως και ελπίζουμε να συνεργαστούμε με όλα τα κράτη-μέλη Ελπίζουμε να υπάρχει συντονισμός με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εφαρμογή όμως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή, μηδενική ανοχή, σε σχέση με την μη μεταγραφή ε, στην εθνική νομοθεσία ε, των ε, αποφάσεων αυτών. Ως πολιτικό όργανο σας ζητώ να συμμετέχετε σε αυτή την σε αυτή, στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής και το λέω αυτό σε σχέση με αυτά που έχει πολλές φορές πει ο κύριος Φαμπ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι μια, ένα εγχείρημα προϋπολογισμού και λογιστικής, ε, το οποίο έγινε ένα οικονομικό εγχείρημα, όχι μόνο όμως στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και σε άλλες επιτροπές. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, το, τη γραμματεία εσένα Μάλκολμ και να μην ξεχάσουμε την ε, ε, ποιότητα και την ειλικρινή δουλειά που μπόρεσα να κάνω μαζί σας ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Well, thank you very Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια εξαιρετική επισκόπηση, κατά την άποψή μου, τονίσατε τα σημαντικότερα θέματα. Και από δική μας πλευράς, και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλων των μελών, όταν λέω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δική σας προσωπική δέσμευση και αφοσίωση σε όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ότι κάθε εισηγητής και ασκιώδης εισηγητής έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή μαζί σας κατά τη διάρκεια της δουλειάς του. Έχετε μια πολύ καλή αίσθηση των πραγμάτων. Ήσασταν και πολύ ανοιχτό στις δικές μας ιδέες. Μιλήσατε για ε, την ε, πράξη για την ενιαία αγορά, που ήταν μια πολύ καλή ιδέα, ε, που προωθήσαμε από κοινού με άλλες ιδέες και σκέφτομαι τον αριθμό των φυλαδίων ε, που έχουμε τώρα στα γραφεία μας. Εκτός από αυτό ε, το φυλάδιο έχουμε και τις 10 ε, κυριότερες ανησυχίες των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν δική μας ιδέα, τι πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το φόρουμ της σειράς Αγοράς και η παρακολούθησή του, η ενέργεια με την οποία δουλέψατε μαζί σας για ε, να ε, καταστεί πιο σημαντική η ενιαία αγορά είναι πραγματικά αξιέπαινη. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι, είναι... έχουν ως αποτέλεσμα αυτήν την ε, ε, δουλειά στην οποία καταλήξαμε και στην οποία ελπίζω να συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία. Γκέπχαρντ, έχω ξεχάσει κανέναν. κυρία Λεγκρίπ και η κυρία Λεγκρίπ νομίζω. Λοιπόν, τρεις ομάδες τριών ομιλητών. Όχι, δύο των τριών και μία τελευταία ομάδα δύο ομιλητών. Αν δεν προσθεθεί κανένας άλλος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε άλλωστε και έξω στο κοκτέιλ. Η Ριγκόιερ Πέρες, Στάιλερ και Κρόιτσμαν, η πρώτη ομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την πολύ καλή εργασία και όπως τονίσατε για το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι καθηκόντα αναλάβετε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στους Ισπανούς. Είναι μια χώρα που ξέρετε πολύ καλά γιατί την επισκεφτήκατε πρόσφατα τρεις, τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει οι εφαρμογές για το υποκείμενο χρέος, για τις διαφορετικές μορφές ε, χρεών και την ε, ιεραρχία τους σε περίπτωση Δεύτερον, η χειραγώγηση του Euribor που οδήγησε σε ζημιέ για όσου είχαν στεγαστικά δάνεια και επίσης για τη μη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσει σε τόσο μεγάλες ε, εταιρείε, οι οποίες είναι κυρίως δημόσιες αλλά τίποτα δεν φτάνει στις μικρομεσαίε και στι οικογένειε αυτών που τι λειτουργούν. Το πρώτο σημείο δεν κατάλαβα το πρώτο θέμα το οποίο θέσατε. Δεν κατάλαβα για ποια δοκιμή μιλήσατε ακριβώ. Μιλούσα για την υποχρέωση όταν κάποιος αγοράζει ε, υποκείμενο χρέος, δεύτερης προτεραιότητος χρέους ή τις λεγόμενες προτιμησιακές μετοχές όπω έγινε στην Ισπανία, το άτομο αυτό θα πρέπει να καταδείξει ότι έχει κάποια γνώση των χρηματοοικονομικών θεμάτων. Οι περισσότεροι που αγόρασαν τέτοιε μετοχέ προτιμησιακέ στη χώρα μου δεν γνωρίζανε καθόλου ότι ουσιαστικά οι τράπεζε οι οποίε είχαν γεμίσει με αυτόν τον τρόπο τα ταμεία του δεν είχαν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο. Αυτό είναι θέμα ικανότητος πληρωμής ή προσυμβατική υποχρέωση και τέτοια, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία ο προεδρος η κυρια σταιντα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την επισκόπησή σας, για την οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε πολλοί ε, συνάδελφοι να προσέξουν καλά για να ξέρουν τι κάναμε τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την καλύτερη προστασία των πολιτών που αναφέρατε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με αυτό που είπατε για τα οικονομικά θέματα, όταν μιλήσατε για παράδειγμα για την αύξηση, την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε οποιοδήποτε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας και να πάει κανείς ε, υπάρχει ε, μία ανακοίνωση που λέει ότι εγγυώνται τις ε, καταθέσεις μέχρι 85.000 λίρες για, για το κάθε καταθέτη. Μερικές φορές εθνικοποιούμε την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλα τα κακά τα στέλνουμε πίσω στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα ως προς αυτό όσον αφορά τις συντάξεις. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτό το νέο συνταξιδοτικό σύστημα γιατί είναι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Ε, ο κόσμος ενδιαφέρεται και ανησυχεί πολύ για τις συντάξεις του. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει ε, σε ξένες χώρες οπότε θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Και θα ήθελα να μας πείτε ε, τι συμβουλές θα μπορούσατε να δώσετε στο διάδοχό σας για καλύτερη συνεργασία, ειδικότερα για τα ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Και ο κύριος Κρόετσμαν, τελευταίος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να, ευχάσω, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Επίτροπο Μπαρνιέ για τα μάση συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Πάντα ένιωσα μεγάλη χαρά όταν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και βρίσκαμε κοινέ ε, λύσεις. Σκέφτομαι επίμαχα θέματα όπως αυτό των συμβάσεων παραχωρήσεων, να μην συμπεριληφθεί η υδροδότηση παραγματικά. χάρη. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην ε, Γερμανία και κράτησε μια πολύ πραγματιστική θέση ο κύριο ε, Επίτροπος που δέχτηκε την εξαίρεση τη υδροδότηση στον σχετικό τρίλογο. Αναφερθήκατε όμως στο θέμα της ε, των τυχηρών παιχνιδιών στο ίντερνετ. Έχουμε πει ότι χωρίς ευρωπαϊκές λύσεις δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, είτε πρόκειται για αυτούς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα παίγνια ουσιαστικά, είτε των νέων και οι απάτες σε αυτά τα παιχνίδια, οι ευκαιρίε για ξέπλυμα χρημάτων μέσω αυτών των παιχνιδιών, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γερμανία αλλάξαμε το καθεστώς. Δεν έχει εφαρμοστεί όμως ακόμα η αντίστοιχη ρύθμιση και η Κομισιόν άφησε στο χρόνο μέχρι τον Ιούλιο του 2014 για να κάνει αυτή την απαραίτητη αλλαγή στην νομοθεσία. Πώς βλέπετε εσείς την πιθανότητα να υπάρξει πλήρης εφαρμογή ακόμα και μετά την ε, πίεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, εφαρμογή έχουμε 40 αιτήσει για τέτοιες ε, λειτουργίες τυχηροπαιχνιδιών στο, ε, στο διαδίκτυο, 20 από τις οποίες έχουν εγκριθεί. Και θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνονται στο μέλλον πιο γρήγορα από την Κομισιόν οι εξετάσει αυτών των περιπτώσεων. Okay. Uh, uh, Μάλιστα, λοιπόν, μπορεί να απαντήσει τώρα ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Να απαντήσω καταρχάς στην κυρία Ριγκογέν Περές, η οποία μας υπενθύμησε τα πολλά προβλήματα, καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο αδικίας, το οποίο έχει εντοπιστεί στη χώρα της, στην Ισπανία, αλλά όχι μόνο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν κανόνες ή επειδή πολλές φορές έχουν γίνει κάποιες λανθασμένες πληρωμές ή δεν υπάρχει απαραίτητη οικονομική εποπτεία δεν αποτελεί άμεση αρμοδιότητα της δικής επιτροπής, πάντως το ζήτημα αυτό θα πρέπει να σας αφορά ως ευρωβουλευτές, τη στιγμή που θα πρέπει να απευθυνθείτε βέβαια στους ψηφοφόρους σας. Το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, συντοποιώντας πραγματικά ότι αυτά υφίστανται για πάρα πολλούς πολίτες, αλλά ότι έχουμε αντλήσει ουσιαστικά τα διδάγματα από την κρίση αυτή. 28 νομοθετικές προτάσεις εγώ υπέβαλα και παρακολούθησα και είναι πάρα πολύ στιμόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι στα πλαίσια των προτάσεων αυτών θέλουμε μια καλύτερη ρύθμιση, μια καλύτερη επιτήρηση και εποπτεία. Είναι ιδανική τώρα η νόμη αυτή, είναι η καλύτερη δυνατή, προφανώς όχι. Προφανώ υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωση, αλλά μη τι άλλο, έχουμε πλέον ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, μια ρυθμιστική αρχιτεκτονική, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα από τα τελευταία κείμενα τα οποία έχω αναλύσει όσον αφορά την διάρθρωση των τραπεζών είναι ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει περισσότερο το επόμενο κοινοβούλιο. Πιστεύω πάντως ότι με τα νομοθετήματα που έχουμε ήδη εγκρίνει έχουμε αντλήσει πλέον τα διδάγματα της Κρήτης και κυρίως κυρία Συρικογέν Περές όσον αφορά το ζήτημα της ενημέρωσης των καταναλωτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε στα ζητήματα της κατάχρησης που είχαμε στην χώρα σας, αλλά με την έγκριση των πρίψ της δέσμης των επενδυτικών προϊόντων και τους ιδιώτες επενδυτές, θεωρώ πραγματικά ότι καταδεικνύουμε ότι έχουμε αντλήσει τα διδάγματα της κρίσης για τις πιο ευάλωτους καταναλωτές. Εγώ θα ήθελα και μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας να έχουμε εγκρίνει το κείμενο για την συγκριτική αξιολόγηση, αλλά όσον αφορά το Eurolibor, το οποίο χρησιμοποιείται στην Ισπανία σε πάρα πολλά σε πάρα πολλές συμβάσεις δανειοδότησης για την αγορά σπιτιών, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πραγματικά σκανδαλώδης. Ξέρετε, όταν μιλούσαμε για το Eurolibor ή για τη συγκριτική αξιολόγηση, είχα πει τότε ότι θα πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να καταστήσουμε πιο αυστηρή την νομοθεσία για την κατάχρηση τη αγορά. Πράγμα το οποίο έγινε και αυτή τη στιγμή μπορούμε πραγματικά να διώξουμε ποινικά του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι παράνομα λειτουργήσαν κατά το Ευρωπαίου πολίτη, κατά του ίδιου του κράτου του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα και ελπίζω το κείμενο για το benchmarking να υιοθετηθεί σύντομα. Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα. Η απάντηση δόθηκε θεωρώ μέσω της Τραπεζικής Ένωσης. Η οικονομική αυτή κρίση όχι μόνο έβαλε κατά της οικονομικής ανάπτυξης προφανώς σε πάρα πολλές χώρες, αλλά παράλληλα εμπόδισε αυτό το οποίο τότε βλέπαμε να αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά την διατραπεζική συνεργασία. Και ανταυτού είδαμε ότι οι τράπεζες οι εθνικές αναδιπλώθηκαν πάλι στον εαυτό τους και σταμάτησαν να δανείζουν η μία στην άλλη. Ο κατακαιρματισμός αυτός είναι κάτι το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα και ένα 83% των γερμανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταφέρει να έχει πρόσβαση σε δανειοδότηση σε, με χαμηλά επιτόκια. Ενώ 45% μόνο των επιχειρήσεων στην Ιταλία και στην Ισπανία, 23% για την Ελλάδα με επιτόκια πολύ πιο υψηλά. Καταλαβαίνετε ότι η άνηση αυτή η εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα λοιπόν από το ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί πάλι η διατραπεζική δανειοδότηση μέσω σημαντικών δανείων είναι πάρα πολύ σημαντικό η όλη αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθεί μέσω της Τραπεζικής Ένωσης. Να έχουμε δηλαδή μια πιο ομοιόμορφη και καλώς λειτουργούσα αγορά τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υπάρχουν πολλά άλλα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέσου αυτού που ελπίζω να ξαναχρησιμοποιήσουμε με ιδιαίτερη όμως προσοχή, με ιδιαίτερη διαφάνεια, το ζήτημα της τιτλοποίησης, το μέσο της τιτλοποίησης. Δεν υπάρχει λόγο να σας πενθυμίσω πραγματικά τις επώδυνες συνέπειες της κακής τιτλοποίησης στις ΗΠΑ. Πάντως θεωρώ ότι προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη γκάμα Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το μέσο τη εκπλοποίηση, αρκεί όμω να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνε. Και υπάρχει και άλλη μια συγκεκριμένη ιδέα, την οποία έθεσα για την ιστορική αγορά, τη δημιουργία ενό αποταμιευτικού λογαριασμού ευρωπαϊκού. Δηλαδή πέρα από του εθνικού ε, τραπεζικού αποταμιευτικού λογαριασμού, θα έχουμε και ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό λογαριασμό, πάλι με συγκεκριμένα πρότυπα, προκειμένου να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε την ανθούσα αποταμίευση που έχουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και να τη διοχετεύσουμε προς τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Η κυρία Στάιλερ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αποταμιεύσεις και ως προς αυτό έχουμε αντλήσει διάφορα διδάγματα. Ο κανόνας όσον αφορά της, ε, η νέα ρύθμιση όσον αφορά τις αποταμιεύσεις ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγγυώνται όλες, εγγυώμεθα όλες τις αποταμιεύσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Εγκρίθηκε λοιπόν ο κανονισμός αυτός προκειμένου πραγματικά να υπάρχει μια ομοιόμορφη κατάσταση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 28 τέτοια αποταμιευτικά ταμεία αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προϊόντος του χρόνου θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα αυτά εθνικά ταμεία, όπως άλλωστε λέγεται και στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ρωτήσατε κυρία Στάιλερ τι συμβουλές θα μπορούσα να δώσω, όχι προφανώς στους ε, νέους ευρωβουλευτές, αλλά τουλάχιστον στον άνθρωπο που θα με διαδεχθεί Αυτό που θα έλεγα είναι ότι όχι μόνο έχουμε τη νέα συνθήκη η οποία ενισχύει τις αρμοδιότητες συναπόφασης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πιο ποιοτικά νομοθετικά κείμενα, πιο εύληπτα τέτοια κείμενα, τα οποία να εξηγούμε καλύτερα προς τα έξω, προς τις εκλογικές σας περιφέρειες, προς τον Ευρωπαίο πολίτη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό ο νέος επίτροπος να μην είναι δύσπιστος απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι πολλές φορές είστε πολύ επικριτικοί είναι δύσκολη πολλές φορές η αντιμετώπιση των δικών σας των επικρίσεων, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μελλοντικός επίτροπος να συνεργαστεί στενά μαζί σας. Αυτή θα είναι η βασική συμβολή που θα του έλεγα. Να συνεργαστεί, να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά όλε αυτέ τι εκθέσει πρωτοβουλία τι οποίε έχετε εσείς και πραγματικά ανοίγουν το δρόμο για μα. Πολύ περισσότερο εφάνταστα είναι και πρωτοποριακά είναι αυτά τα κείμενα από ό,τι θα μπορούσε να κάνει να συντάξει ένας υπάλληλο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην νομοθεσία την οποία εγκρίνουμε. Πρέπει να ισχύουν οι συνθήκε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και να δείξουμε μηδενική ανοχή. Παράλληλα όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα ανάμεσα στους νομοθέτες. Αυτό προσπάθησα εγώ να κάνω σε όλους αυτούς τους τριμερείς διαλόγους που είχαμε. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια στρατηγική. Και συνεργαζόμενος με τον κύριο Ταγιάννη ασχολήθηκα και με το ζήτημα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσει μια στρατηγική βιομηχανικής ανταγωνιστικότητος. Ήμασταν ιδιαίτερα θαραλέοι με την κοινή γεωρική πολιτική πριν από κάποια χρόνια. Για ποιο λόγο να μην δείξουμε το ίδιο θάρρο για μια στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε κοινέ επενδύσει με συμμετοχή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στους τομεί εκείνους όπου γνωρίζουμε ότι πραγματικά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό δυναμικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα 20-30 χρόνια. Για ποιο λόγο να χάσουμε τις ευκαιρίε αυτές, για ποιο το λόγο τις επενδύσεις αυτές να τις κάνουν τελικά άλλοι, οι Αμερικάνοι ή οι Κινέζοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε κοινέ επενδύσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για κάποιους βασικούς βιομηχανικούς τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι αυτή η οποία θα πρέπει με τη δική σας συνεργασία να κάνει μια τέτοια πρόταση για τη βιομηχανική στρατηγική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κρόιτσμαν για την εργασία την οποία έκανε στα πλαίσια των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωσή μα το 2012 είχα πει ότι έχουμε 15.000 ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με τυχερά παιχνίδια, εκ των οποίων άνω το 85% λειτουργούν χωρίς άδεια, ουσιαστικά λειτουργούν παράνομα. Εσείς τότε Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη θεσμική συνεργασία προκειμένου να προστατευτεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής και μας είχατε πει ότι θα πρέπει να διευρύνουμε περισσότερο την νόμιμη προσφορά των παιχνιδιών αυτών και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την πειρατεία. Κατά πολέμηση πειρατείας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στραφούμε κατά των νέων αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πειρατικά αυτά παιχνίδια. Αντίθετα, θα πρέπει να τους προσφέρουμε μια καλύτερη και μεγαλύτερη νόμιμη αγορά τέτοιων παιχνιδιών και να τους ενημερώσουμε για το κόστος που έχει η πειρατεία όσον αφορά την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό καταφέραμε να προσφέρουμε κάποιες, κάποια νόμιμα τυχερά παιχνίδια και Προσπάθησα πραγματικά να ευνοήσω τις νέες αυτές ευκαιρίες παρά να επιβάλλω κάποιους περιορισμούς, αλλά νομίζω ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί και θα χρειαστούμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα τυχερά πνεχνίδια, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα της απάτης και όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια στον τομέα του αθλητισμού και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε επίσης και τους ανήλικους. Θα έλεγα λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι θα με διαδεχθούν ότι εγώ προσπάθησα να προωθήσω τις ε, νόμιμες αν θέλετε προσφορές ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιους κανόνες. Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές πίσω από τα παράνομα τυχερά παιχνίδια κρύβονται ε, εγκληματικές οργανώσεις, κρύβεται η μαφία. Μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία παρανόμως νομιμοποιούνται μέσω των παιχνιδιών αυτών. Είτε μιλάμε λοιπόν για τα τυχερά αυτά παιχνίδια και τη νέα αυτή αγορά, είτε μιλάμε για την παράνομη αυτή, τα παράνομα παιχνίδια, χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ένα νέο νομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε, για τις ε, απαντήσεις σας και τα επόμενα τρία ερωτήματα από την Τεπανιό, τον ε, Άντρε Σουάπ και την Χάιντι Ρούλε. Σε ευχαριστώ. Μάλκολμ, σήμερα Νομίζω ότι φυσικά είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας, τελευταία μας συνάντηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Κύριε Επίτροπε, τελικά κάνατε ένα απολογισμό ουσιαστικά εξαντλητικό όλων αυτών που πετύχαμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια μαζί, εγώ από τη δική μου πλευρά, αλλά νομίζω ότι είναι και η κοινή αντίληψη. Εργαστήκαμε πραγματικά πολύ θετικά μαζί σας, υπηρετώντα το γενικό, το συλλογικό μας συμφέρον, και πέρα από τις διαφορές που μπορεί να είχαμε, πέρα και από τις θεσμικές διαφορές που μπορεί να υπήρξαν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά για να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον. μια μεγάλη χαρά για όλους μας να εργαστούμε και ως Κοινοβούλιο και μαζί σας. Ποτέ δεν νομίζω ότι είχαμε κάνει τόσα πολλά πράγματα προς την κατεύθυνση του κοινού συμφέροντος και για να αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές και τους πολίτες είναι γεγονός ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε μια κόποση σε σχέση με την εσωτερική αγορά και αυτή την κάποια αποστροφή που ένιωσαν ακόμα οι πολίτες για την ενιαία αγορά. Αυτό ήταν η μόνη μας μέρημνα στη συνεργασία μαζί σας και αν είχα τώρα να διατυπώσω ε, μια ευχή για τα επόμενα χρόνια θα ήταν να υπάρξουν πολλοί επίτροποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με το σύνολο όλων αυτών των θεμάτων και όλες οι υπηρεσίες τους στα πλαίσια της Κομισιόν, γιατί έχω εργαστεί όχι μόνο μαζί σας αλλά και με τις υπηρεσίες σας και θέλω να πω ότι σοφόρα τιμής, ήταν όλα αυτά πολύ θετικά και ελπίζω να γίνουν και στο μέλλον, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε τις μεθόδους εργασίας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε πιο αγαπητή την ενία αγορά στους πολίτες, φυσικά έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά εγχειρήματα να φέρουμε σε πέρας, όπως είπατε, υπάρχει πολλές φορές ο κίνδυνος, ο μεγάλος κίνδυνος που προέρχεται από τη μακρά διαδικασία μεταγραφής στο εθνικό δίκαιο που πολλές φορές προσκρούει σε αμφισβητήσεις και μπορεί να αλλοιώσει την αρχική μας πρόθεση αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι οι δικές σας υπηρεσίες οι οποίες παραμένουν πάντα, εμείς δεν έχουμε τέτοια μονιμότητα, δεν είμαστε πάντα παρόντες, θα πρέπει οι υπηρεσίες της Κομισιόν να δείξουν μεγάλη επαγρύπνηση και να εξασφαλίσουν ότι μεταξύ και των μελών του Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Συμβουλίου και των βουλευτών και των συνεργατών τους θα υπάρξει και στο μέλλον μια αντίστοιχη σύμπνοια σε σχέση με την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Η ιδέα που ξεκινήσατε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο Αποταμίευσης μπορεί και αυτή να συμπληρώσει όλα αυτά που έχουμε κάνει για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια δημιουργήσαμε από κοινού εργαλεία ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά αυτό το βιβλιάριο αποταμίευσης θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της καινοτομίας, της έρευνας που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης και επίσης το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που αναφέρθηκε ή δεν αναφέρθηκε, θα πρέπει και αυτό να μπορέσει να ευδοκιμήσει είναι πολλά αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Πολλές φορές η πρακτική εφαρμογή δεν ήταν πάντα εύκολη. Γι' αυτό βασίζομαι σε αυτούς που θα παραμείνουν στην Επιτροπή μας και τους νέους συναδέλφους και τις υπηρεσίες της Κομισιόν για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ξεπεράσουν τις πολιτιστικές και πολιτισμικές διαφορές που έχουμε μεταξύ των χωρών μας και να προχωρήσουμε αυτά που ξεκίνησαν αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο Άντερ Φαμπ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μισελ Μπαρνιέ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, για το σημαντικό έργο που έκανες και από την Επιτροπή μας και από τους βουλευτές του ΕΛΚ θέλω να σε ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την καταπληκτική αυτή συνεργασία που είχαμε. Είναι φανερό ότι πετύχαμε πολλά πράγματα και αυτό αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και για μένα υπήρξαν οι πιο σημαντικές πρόοδοι στα θέματα της, της ε, εσωτερικής αγοράς και είναι δυτή αυτή η πρόοδος. Πρώτα απ' όλα με την νομοθεσία για την ενιαία αγορά μπορέσαμε και πάλι να έχουμε μια οριζόντια εναρμόνιση για διάφορα τμήματα της εσωτερικής αγοράς και εξασφαλίσαμε και μια σωστή εναρμόνιση των προσπαθειών μέσα στην υπηρεσία της Κομισιόν, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν είχε επιτευχθεί αυτό τόσο πολύ. Όλα αυτά εξασφαλίστηκαν με την ε, νομοθεσία για την αγορά, το Single Market Art και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα μπορέσει να υπάρξει η σωστή συνεργασία των επιτρόπων για μια κοινή πολιτική στην εσωτερική αγορά. Αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο. Δεύτερον, έχω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έννοια της μηδενικής ανοχής που ανέφερες. Ξέρω ότι η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και ο καλύτερος έλεγχος αυτού που κάνουν τα εθνικά κράτη για αυτό που αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να αντιμετωπίσετε μονάχα με μηδενική ανοχή, αλλά και με μια κοινή στρατηγία ώστε η Κομισιόν να μπορεί να εξασφαλίζει ότι λειτουργεί σωστά η εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων στα κράτη-μέλη σε ένα ομοσπονδιακό σχήμα χρειάζονται και τα κράτη-μέλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τούμπαλη. Και πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια επαγρύπνηση για να ισχύει αυτό το θέμα. Και φυσικά, εάν δεν θέλουμε να αφήσουμε να μας κυριεύσει ο λαϊκισμός, είναι απαραίτητα όλα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Και θέλω να σταθώ τώρα σε μερικά, σε δύο σημαντικά ε, θέματα. Πρώτο το θέμα των ρυθμιζομένων επαγγελμάτων και τι θέλει να κάνει η Κομισιόν για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα είναι πιο ανοιχτή η ευρωπαϊκή αγορά για αυτά τα επαγγέλματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι και επίση υπάρχει και έλλειψη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Γι' αυτό θέλω να θέσω το συγκεκριμένο μου ερώτημα πώς πάνε τα πράγματα με την επεξεργασία της ε, αλλαγής των ε, εθνικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση στα επαγγέλματα, αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χάρτης για την πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα, ώστε να έχουμε την ελπίδα ότι κάπου θα υπηρεπιδηθούν όλα αυτά τα εμπόδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άντες, η Χάιντι Ρούλια και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Επίτροπο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μαζί σας και φυσικά και την γραμματεία σας, τους συνεργάτες σας, τους δικούς μας συνεργάτες και θέλω φυσικά να, εφαρμο... να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάλκομ Χάρμπορ, εξ ονόματο τη ομάδα των Πλασίλων, γιατί την είχα προηγουμένω την ευκαιρία αυτή. Είναι η τελευταία μα συνεδρίαση, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα σαφέ ότι ήταν πολύ θετικά αυτά τα πέντε χρόνια, ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μα και μεταξύ μα και με τον κύριο Επίτροπο. Αυτό όμως έγινε πραγματικά όταν και ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του στην Επιτροπή μας παίζουν και αυτοί το ρόλο τους. <clears throat> Θέλω επίση να σας τονίσω και τις ευχαριστίες των Δήμων και Κοινοτήτων της, ε, από την Αυστρία με τους οποίους μίλησα για τα θέματα των συμβάσεων παραχώρησης. Υπήρξε πραγματικά μια ικανοποίηση για το γεγονό ότι αυτή η οδηγία μπόρεσε να προχωρήσει φέρνοντα μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και ασφάλεια δικαίου και απλοποίηση και είναι κάτι το οποίο οφείλεται και στι δικέ σα προσπάθειε. Θέλω να έρθω στο δεύτερο ζήτημα που αναφέρατε εσεί, το θέμα τη εφαρμογή, τη μεταγραφή και εφαρμογή των νομοθετημάτων σε πολλού τομεί. Όπω παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να θέσουμε σε, στο προσκήνιο τον έλεγχο της ε, εφαρμογής τους και να μην προχωρούμε τόσο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις. Γιατί για το θέμα αυτό των, της αμοιβαία αναγνώρισης των ε, ε, προσόντων είδα ότι υπήρξαν τρεις μεταρρυθμίσεις στο χρόνο που ήμουν στο Κοινοβούλιο και αυτό μου φαίνεται υπερβολικό. Πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε και το ερώτημα με ποιο τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη βιομηχανική πολιτική η οποία θα υποστηρίξει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη νομοθεσία η οποία να έχει μια κάποια χρονική διάρκεια και η οποία δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τη δική σα υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί η διάρκεια τη νομοθεσία στον τομέα αυτό. Μήπως ε, η κυρία Λεγκρίπ ε, και η κυρία Γκέπχαρτ ε, θα μπορούσαν να ρωτήσουν τώρα, να κάνουν τώρα τις ερωτήσεις τους. Μπορώ να συνεχίσω ακριβώς εκεί που σταμάτησε η προελαλή σας. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα κύριε Επίτροπε Μπαρνιέ για την πολύ καλή συνεργασία, το ανοιχτό πνεύμα το οποίο υπήρξε στη συνεργασία μεταξύ μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε για όλους τους επιτρόπους δυστυχώς και στα 20 χρόνια που έχω βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω ζήσει πολλές εμπειρίες που δεν ήταν τόσο θετικές. θετικές. Και θα έπρεπε κι εσείς να θυμίσετε στους ε, ε, διαδόχους ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και το ανοιχτό πνεύμα, η διαδικασία συνεργασίας και το ανοιχτό πνεύμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι θεμελιώδες. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη είναι το γεγονός ότι υπάρχουν με μεγάλη ε, ταχύτητα αλλαγές μέσα στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραγωγή, χάρη το θέμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Εμείς είπαμε δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτή την οδηγία. Πρέπει πρώτα όμως να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται η εφαρμογή και να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται σωστά η εφαρμογή των κανόνων για τις συμβάσει, για ε, υπηρεσίε, συγγνώμη. Να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη σταθερότητα και ε, εμπιστοσύνη για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με το να μην αλλάζουν συνέχεια οι κανόνες. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσετε ότι θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι κανόνες και να καταλάβουμε την ελεπίδραση αυτών των κανόνων με τους άλλους νομικούς κανόνες προτού προχωρήσουμε σε νέα κείμενα και νέες προτάσεις. Και κυρίως προτού υπάρξει η πλήρης εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Ευχαριστώ πολύ και η κυρία Λεγκρίπ τελευταία ομιλήτρια για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, συγγνώμη αν ε, και εγώ επαναλαμβάνω τα ίδια μετά από τους προλαλήσαντες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ποιότητα της εργασίας ε, που ολοκληρώσαμε μαζί και για, την, ε, το γεγονός ότι πάντοτε μας ακούγατε, πάντοτε ήσασταν διαθέσιμος, πάντοτε έρχεστε να μας δείτε στο Κοινοβούλιο και ειδικότερα εμάς στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ελπίζουμε ότι αυτή η πολιτική θα ε, συνεχίσει ε, και θα εμπνεύσει και τα μελλοντικά μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Θα ήθελα να σας επενέσω εσάς και την ομάδα σας, ε, τους συνεργάτες σας, ε, γιατί η εσωτερική αγορά αποτελεί και πάλι επίκεντρο ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής γιατί αποτελεί θεμέλιο λίθο της δικής μας δουλειάς και είναι ο λίθος πάνω στον οποίο θα οικοδομήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω ερωτήσεις, απλώς να εκφράσω αυτήν την ε, επιθυμία, τη δική μου, είναι λίγο ιδιαίτερη η θέση μου στην Επιτροπή Εσωτερικών ε, Θεμάτων. Μετά από την ανάληψη των καθηκόντων σας, ε, εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Ένα μικρό λοιπόν προσωπικό σχόλιο. Νομίζω ότι στο μέλλον, στα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό προσδοκούν ε, οι πολίτες μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εργαστούμε ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο απλοί, να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή η νομοθεσία, ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να υπάρχει και σταθερότητα ε, νομική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας από, τους, από τις βασικές προσδοκίες. Πρέπει βέβαια να ολοκληρώσουμε και την δουλειά της ε, εσωτερικής αγοράς, ε, αλλά πρέπει παράλληλα να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη αυτή για σταθερότητα ε, της, ε, των, της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να μας πει κάποια καταληκτικά σχόλια και να απαντήσει ερωτήσεις. Με πολύ χαρά έγινα μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2010 και με αντικατέστησε η συνάδελφος για να απαντήσω στην Περναντέτ Βερνιό, την οποία θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω, αλλά και την κυρία Γκέπχαρτ και την κυρία Ρούλε. όλοι σας και οι Κωνστόνς μιλήσατε για την εφαρμογή των ε, κειμένων. Οπότε καλό θα ήταν να πω ορισμένα πράγματα. Λίγα περισσότερα πράγματα λοιπόν για τη μηδενική ανοχή της μη μεταγραφής ε, της νομοθεσίας, ε, που την υπογραμμίζω και πάλι. Στην, βλέπουμε ότι μόνο δύο κράτη-μέλη ε, η Πολωνία και το Βέλγιο δεν έχουν καταφέρει να ε, επιτύχουν το στόχο του 1% ακόμη. 0,6 είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα θέλουμε να πάμε και στο 0,5 το οποίο προτείναμε στην πράξη για την ενιαία αγορά και είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Μου φαίνεται ότι είναι ένας από τους φιλόδοξους και απαιτητικούς στόχους που για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια ε, εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί στο 100% της. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό που μας είπατε. Το ελάχιστο λοιπόν ιστορικό η απάντησή μου αφορά το scoreboard το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ε, η κυρία ε, Βέρνιο. Ελπίζω μετά από το 0,5 να πάμε ακόμη και πιο κάτω. Υπάρχει πρόοδος βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, τώρα, το θέμα της ε, αμοιβαίας αξιολόγησης και το εγχείρημα αυτό. Πρέπει να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν για την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλματα ε, είναι σορευτικές, ε, συχνά οι περιορισμοί για την πρόσβαση σε ένα, ε, σε ένα επάγγελμα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε ήδη δει από την παρουσίαση, στην παρουσίαση της πρότασής μας για, την, για τις υπηρεσίες. Θέλουμε να δώσουμε μία ε, πλήρη διαφάνεια στους επαγγελματίες, ειδικότερα ε, στα κράτη-μέλη όπου χρειάζονται συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Νομίζω λοιπόν η συγκρισιμότητα και η διαφάνεια θα, είναι ένα, θα, θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ώστε κάποια εμπόδια που έχουν μόνο προστατευτικό χαρακτήρα να μπορούν να ε, απομακρυνθούν ευκολότερα αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα εξυγχρονισμό της νομοθεσίας ε, για τα επαγγέλματα στα κράτη-μέλη και θα καλέσουμε κάθε κράτος μέλος ε, να εξετάσει τους ε, περιορισμούς πρόσβασης στα επαγγέλματα και νομίζω ότι σε αυτήν την αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αλλά στους επόμενους μήνες θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για την ανάλυση μας αυτής αναχώρα. σε σχέση πάντοτε με τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Η οριζόντια ε, διαβούλευση, η μέθοδος αυτή της ε, ε, βαθμολόγησης σε σχέση με τα εμπόδια και αυτή η αμοιβαία ενημέρωση θα είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορεί το επόμενο κοινοβούλιο να το χρησιμοποιήσει ως γνώμονα για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ρούλε για την αξιολόγησή της. Ο στόχος ήταν να μειώσουμε τους περιορισμούς. Εγώ ήμουν πρόεδρος μιας ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, για 20 χρόνια περίπου και είδα πώς ε, απέτρεπαν ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ορισμένα μέτρα γιατί τους στήχησε το 30% του τζίρου τους. Οπότε επανέρχομαι και στο θέμα της καινοτομίας, είναι κάτι για το οποίο με είχε ρωτήσει ο Μάλκολμ. Η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, όλα αυτά πρέπει να ε, εξασφαλιστούν νομικά. Εύελιν Γκέπχαρτ σημείωσε αυτό που είπατε για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μία μεταγραφή σωστά, πρέπει να γνωρίζουμε το τελικό νομοθετικό κείμενο. Όταν βλέπουμε τι γίνεται, για παράδειγμα, με τις δημόσιες συμβάσεις ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε μια αξιολόγηση προτού ε, να γνωρίζουμε το νομοθετικό κείμενο, το οποίο συχνά διαφέρει κατά πολύ από την αρχική πρόταση. Εγώ βέβαια παίρνω πολύ σοβαρά όλες αυτή, όλη αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου τα σχετικά κείμενα. Αυτό που κάναμε με ε, τους τοπικά ε, εκλεγμένους, με τους stakeholders, εμπλεκόμενους, είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπατε και για την εκτίμησή σας και να επανέλθω σε αυτά που είπε η Constance Grip για την εσωτερική αγορά που είναι η βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η οικονομική κρίση κατέστησε την εσωτερική αγορά το πρώτο ενδεχόμενο θύμα αυτής της ε, κρίσης γιατί πριν, ε, ε, γιατί υπάρχει ο εθνικισμός, υπάρχει ο προστατευτισμός και υπάρχει και η αποδόμηση της εσωτερικής αγοράς. Επομένως, αν δουλεύει καλύτερα η εσωτερική αγορά, μπορούμε να βρούμε κάποια σημεία ανάπτυξης ε, και μιλάω ας πούμε για τις ε, συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς να διευκολύνουμε τις συναλλαγές και γι' αυτό ακριβώς εγώ αφοσιώθηκα με όλους τους συνεργάτες μου ε, στην προσπάθεια αυτή να είναι κάπως πιο πραγματική η προσέγγιση ε, και για τους ε, πολίτες δεν ε, είναι θέμα ματαιοδοξίας. Ε, είναι πάρα πολύ λογικό να αξιολογούμε αυτά που καταφέραμε να πετύχουμε μαζί, αλλά ας μην εφησυχάζουμε γιατί υπάρχει πολλή ανεργία, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για να ε, εφησυχάζουμε υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η Ευρώπη είναι χρήσιμη, ότι δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ε, ζωής μας και ότι επιφέρει πρόοδο και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο πρέπει να το, να χρησιμοποιήσετε στον, ε, στις προεκλογικές σας εκστρατείες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την νομική υπηρεσία της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όλους τους συνεργάτες μου κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μισελ Μπαρνιέ, σε ευχαριστούμε πραγματικά γιατί ολοκληρώνουμε μαζί με ένα τόσο δυναμικό τρόπο και προορατικό τρόπο την πενταετή μας αυτή θητεία. Ξέρω ότι πραγματικά σε άκουσαν πάρα πολύ προσεκτικά, οι οι βουλευτέ αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν και στο επόμενο κοινοβούλιο. Έχουμε, μάλλον, έχουμε καθυστερήσει κατά ένα λεπτό. Θα ήθελα απλώ να μιλήσω και εγώ λίγο στα τελευταία αυτά λεπτά, να σα πω κάποιε δικέ μου προσωπικέ απόψει. Όλους ιδιαίτερω θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς ε, συνεργάτες μου, αλλά ενθαρρύνομαι πραγματικά από τα όσα είπατε, από τον τρόπο που πραγματικά προσεγγίζετε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, οι δημόσιες συμβάσει, Πριν από λίγο μιλήσαμε για τον νοσιακό του ελληνικό κώδικα. Ε, πρέπει επίση να συζητήσουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πρότυπα για τι επιχειρήσει. Ε, δεν ακούσαμε βέβαια σήμερα τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Θυμάστε ότι αρχικά εγώ, σε συνεργασία με τους συντονιστές καταφέραμε να εργαστούμε πολύ επικοδομητικά και να τους ευχαριστήσω γιατί αυτοί όντως συμβάλλουν στην επικοδομητική συνεργασία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Από κοινού καταφέραμε να αποφασίσουμε για τη στρατηγική που θα ακολουθούσαμε, από κοινού καταφέραμε να προετοιμαστούμε για τον, την άφηξη των νέων αυτών κειμένων και προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εργασία αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω και το εύχομαι ότι η νέα Επιτροπή ΕΜΚΟ αλλά και οι υπόλοιπε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αρχίσουν να λειτουργούν και αυτέ κατά τρόπο. Θεωρώ ότι ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή καταδείξαμε ότι μπορεί κανεί με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσω επικοδοματική συνεργασία να αντιμετωπίζει πολύπλοκα θέματα όπω αυτά τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη δική μα την Επιτροπή. Βέβαια, πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια κρύβεται μια τεράστια προσπάθεια να ευχαριστήσω τον Πάνο και την ομάδα του και τον Τζόρνταν, ο οποίο ήταν ο προκάτοχό του, και να ευχαριστήσω και όλη τη γραμματεία τη Επιτροπή μα η οποία πραγματικά έχει πάρα πολλές καλές ικανότητες και ήταν ιδιαίτερη χαρά το ότι συνεργάστηκα μαζί τους. Να ευχαριστήσω βέβαια και όλα τα μέλη της Επιτροπής, καθώς επίσης και τους συμβούλους από τις πολιτικές ομάδες, οι οποίοι είναι πάντα παρόντες εδώ στα δεξιά μου, και να ευχαριστήσω επίσης και τους βοηθούς των Ευρωβουλευτών, γιατί και αυτοί συμβάλλουν πάρα πολύ στην κοινή μας συνεργασία. Να ευχαριστήσω προφανώς και εσάς και τη δική σας την ομάδα και όλους τους ευρωβουλευτές, όλους τους συναδέλφους μου. Πραγματικά ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά να εγούμε μια τέτοια ταλαντούχα, ενδιαφέρουσα ομάδα ανθρώπων και ήταν πραγματική τιμή για μένα το να μπορώ να ηγούμε αυτή τη επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτές ήταν οι τελευταίες μου παρατηρήσεις. Θα πιούμε τώρα και ένα ποτό και ελπίζω κύριε Επίτροπε να πίνετε κι εσείς λίγο μαζί μας για να πιούμε μαζί ένα ποτό. Ολοκληρώνοντας, ως συνήθω, θα ήθελα να σας πω ότι πρώτον πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Θεωρώ ότι τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια μια σημαντική καινοτομία ήταν ότι όλες μας οι συνεδριάσεις μεταδόθηκαν μέσω του διαδικτύου. Εργαστήκαμε σκληρά και ξέρουμε ότι υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα κρατήριο. και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλου μα ακούνε ακόμα από το διαδίκτυο ότι μπορείτε να λάβετε αυτό το περίφημο ενημερωτικό μα φυλάδιο, το newsletter, αν μα στείλετε ένα απλό email. Δεν ξέρω πόσους συνδρομητές έχουμε, 2.500 νομίζω. Έχει κανείς τον συγκεκριμένο αριθμό, 2.500 συνδρομητές, καταπληκτικά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε μόνο με 200-300 συνδρομητές και φτάσαμε στους 2.500. Αυτό καταδεικνύει το ευρύτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για την Επιτροπή μας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Πρόκειται για την συνεδρίαση σύνθεση σε σώμα που θα εκλεγεί ο νέο πρόεδρο και τα νέα μέλη τη Επιτροπή. Ξέρω όμω ότι πολλοί από εσά θα εξακολουθήσουν να είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ω συνήθω να ευχαριστήσω και του δερμηνεί μα, οι οποίοι κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά και νομίζω, λέει ο πρόεδρο, ότι μπορούμε να του χειροκροτήσουμε. Uh, Ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίαση και καλώ και τους διερμηνείς να έρθουν για ένα ποτό εκτός αιθούσης. Υπάρχει ένα μικρό μπαρ το οποίο έχουμε στήσει έξω από την αίθουσα και μπορούμε εκεί πέρα να πιούμε ένα ποτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. για τη συνεδρίαση.